διάταξη για τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτο 2016 και θα ήθελα εξ αρχή να επισημάνω το εξή, ότι δεν θα έχουμε τη δικασία Catch the Eye και ούτε γαλάζιε κάρτε ε, στην ε, συζήτηση αυτή γιατί η συμφωνία είναι ένα ομιλητή ανά ομάδα. Καταρχά όμω, το λόγο έχει ο Φραντ Τίμερμαντ, ο πρώτο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς πριν από 10 χρόνια στο Λονδίνο πέθαναν 52 άνθρωποι και είχαμε εκατοντάδες ε, τραυματίες σε μια τρομακτική τρομοκρατική επίθεση. Θυμάμαι ζωντανά αυτές τις ημέρες, θυμάμαι την ε, ε, τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης όχι μόνο στο Λονδίνο και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το περιστατικό στην αρχή της παρουσίασής μου διότι πιστεύω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι όποια θέση και αν έχουμε υιοθετήσει για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εκείνη ακριβώς τη στιγμή είχαμε μια αίσθηση κοινού πεπρωμένου. Διότι ό,τι και να κάνουμε, λάθος ή σωστό, έχουμε ένα κοινό καθήκον να αγωνιζόμαστε για το συμφέρον και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Κοινό καθήκον να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι βάρβαροι, αυτοί, αυτοί οι διαταραγμένοι, αυτοί οι μηδενιστές δεν θα είναι σε θέση να φέρουν την καταστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κοινή πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλα τα έθνη που συναποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, είναι πέραν κάθε πολιτικής ιδεολογίας, ε, πέραν ε, κάθε θεωρίας. Είδαμε φοβερέ προκλήσει τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρομοκρατία, η κρίση με τα μεταναστευτικά ρεύματα, η ανάγκη να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία ε, για να αντιμετωπίσουμε τι εξελίξει ε, στην παγκόσμια οικονομία, η Ελλάδα. Αυτό είναι το σκηνικό στο οποίο καλούμαστε εμείς να συντάξουμε το πρόγραμμα εργασίας για το τρέχον και το επόμενο έτος. Θα ήθελα λοιπόν να σας μιλήσω για τα πεπραγμένα μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα εργασίας 2015. Πάνω από το ίμιση του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί σχεδόν 100% χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις άρχισε να είναι λειτουργικό από την 1η Ιουλίου. Έχουμε στρατηγικό θεματολόγιο για τις επενδύσεις, για την Ενεργειακή Ένωση, για την ψηφιακή αγορά, τη μετανάστευση, στην εσωτερική ασφάλεια και ένα δικαιότερο σύστημα εταιρικού φόρου. Αυτά τα προγράμματα εργασίας και τα θεμετολόγια οδήγησαν σε θα οδηγήσουν μάλλον σε ισχυρό νομοθετικό άχθος ε, για τα επόμενα χρόνια. Έχουν φτάσει ήδη κάποιες προτάσεις ε, και άλλες έπονται με την αναθεώρηση για το σύστημα δικαιο... Ε, εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ε, και για την Ενεργειακή Ένωση. Πάνω από 40 προτάσεις απορρέουν από αυτές τις ε, στρατηγικές που έχουμε ήδη καταρτήσει ε, επιπροσθέτω σε σχέση με τις 140 προτάσεις που υπάρχουν ήδη στο τραπέζι των συνονομοθετών. Οπότε ας διαρρήξουμε αυτόν τον μύθο ότι δεν δραστηριοποιείται και δεν ενεργοποιείται αρκετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για θα λειτουργήσουμε σε μεγάλη κλίμακα όταν είναι σημαντικά και μεγάλα τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Φιλόδοξες στρατηγικές ε, για το εμπόριο, για τις επενδύσεις, ε, για τις ε, υπηρεσίες, για την κυκλική οικονομία, πρόγραμμα δράσης, για την δημιουργία μιας ουσιαστικής κεφαλαιακής ένωσης και οι πρώτες νομοθετικές προτάσεις ε, ακολουθούν για τα πιο επίγοντα ζητήματα και πριν το πέρασε το 2015 ε, θα καταθέσουμε ένα ε, ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ΟΝΕ, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Η κοινωνική διάσταση της ΩΝΕ είναι ένα θέμα ε, το οποίο ενδιαφέρει όλος ιδιαίτερος ε, τον κύριο Γιούνκερ και τον υποφαινόμενο. Επίσης, ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα καταστούν διαθέσιμα μέχρι το τέλος του 2015 για την εγγύηση για τους νέους. Επίσης, πακέτο για την ε, κινητικότητα στην εργασία και αυτό θα υιοθετηθεί αργότερα το 2015. Θα γίνουν συζητήσεις επίσης για τις κοινωνικές πολιτικές αμέσως μετά τις θερινές διακοπές. Πρωτού περάσουμε στο 2016, θα ήθελα να τονίσω ότι ε, χρειαζόμαστε τρεις για να χορέψουμε τάγκο ε, παραδόξως πως ε, τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κοινή ευθύνη και γι' αυτό τώρα διαπραγματευόμαστε μια αναθεωρημένη διαθεσμική διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία και προσβλέπω στην πρώτη μας σύσκεψη σε πολιτικό επίπεδο με τον κύριο Σμίτα από την πλευρά της Προεδρίας και με τον κύριο Φερχόφστατ από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσα σε αυτή την πρόταση τονίζουμε την ανάγκη να ολοκληρωθεί το ο ετήσιος και ο πολυετής προγραμματισμός ε, έχοντας ειδικές ρυθμίσεις για τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κοινοβούλιο που αναφέρονται μέσα στη Συμφωνία Πλαίσιο που ήδη τηρούμε και θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε και τηρώντας επίσης ε, το ρόλο που αναλογεί σε κάθε θεσμικό όργανο βάσει των συνθήκων. Ε, λειτουργώντας ανάντι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία μπορούμε με κοινέ προσπάθειες να έχουμε αναβαθμισ συντονισμένα ε, και κοινά αποτελέσματα αντιμετωπίζοντας τις κοινέ προκλήσεις ε, που έχουμε μπροστά μας θα γίνει μία πρώτη συζήτηση προσανατολισμού για το 2016 στο Σώμα των Επιτρόπων. Τώρα, το Σεπτέμβρη θα γίνει ένας απολογισμός για την πρώτη που έχει σημειωθεί και τις μελλοντικέ προκλήσεις στην ετήσια ομιλία για τα πεπραγμένα του κυρίου Γιούνκερ. Για το πρόγραμμα εργασίας του 2016 αναμένεται η έγκρισή του στις 27 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει εντατικό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει φυσικά τη συμφωνίας πλαίσιο και ε, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων θα διαβουλευτεί με τα κράτη-μέλη. Για να υπάρχει μια κατευθυνόμενη συζήτηση θα έχουμε μια επιστολή ε, προθέσεων ε, το Σεπτέμβριο. ταυτόχρονα με το, τη βασική ομιλία του κυρίου Γιούνκερ το Σεπτέμβρη εδώ στο Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε ένα εξισορροπημένο πρόγραμμα εργασίας. Για το 2016 και το 2016 και μόνο θα βασιστούμε και πάλι στις 10 προτεραιότητες που συμφώνησε ο κ. Γιόνκερ με το Κοινοβούλιο. Τα στρατηγικά θεματολογία που ήδη έχουμε παρουσιάσει και αυτά που αναμένονται μέχρι το πέρας του 2015 ε, ε, εξυπακούτο θα είναι το βασικό μας πλαίσιο διατηρώντας έτσι μια εστίαση σε αυτά που έχουμε ήδη προανακοινώσει. Οπότε σας παρακαλώ να θυμάστε θυμάστε πως Αυτά είναι τα κομβικά σημεία του προγράμματος εργασίας μας. Το ξέρετε αυτό. Ξέρετε ότι αυτό είναι το έρισμα των συγκεκριμένων προτάσεων που θα καταθέσουμε στη συνέχεια και το 2016 φυσικά θα έχουμε και την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και θα είναι μεγάλη πρόκληση για, τα, για το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για το REFIT επίσης θα εστιάσουμε σε αυτό διότι για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις χρειάζεται διαρκή σε προσπάθεια και αν χρειάζεται να ανακαλέψουμε ή να αποσύρουμε ή να αναθεωρήσουμε τις προτάσεις για να εγκριθούν άλλες. Θα τις χαρακτηρίσουμε ως τέτοιες στα πλαίσια του refit. Θα πρέπει να προσανατολισόμαστε βάσει των αποτελεσμάτων που θέλουμε να πετύχουμε και να είμαστε ρεαλιστές εάν χρειάζεται επίσπευση σε κάποιες άλλες διαδικασίες, το ίδιο θα κάνουμε. Θα χαρακτηριστούν ως προτάσεις ρίφιτ και νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες. Εν κατακλείδη. Ε, η ευθυγράμμιση του σχεδιασμού, Πρόεδρε, μπορούν, μπορεί να κάνει τη διαφορά, διότι οι πολίτες ε, θα θεωρήσουν έτσι ότι αυτό είναι τμήμα της λύσης ε, για τα προβλήματα που αντιμετωπίσουν και όχι ένα ακόμη πρόβλημα. αργότερα αυτή την εβδομάδα θα εγκριθεί ένα ψήφισμα στο Κοινοβούλιο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στις προϊούσες συζητήσεις και προβληματισμό μας. Ας συνεργαστούμε, διότι έχουμε αναρρύθμιτες προκλήσεις, περιμένουν πάρα πολλές προσδοκίες οι πολίτες από εμάς, ας δουλέψουμε μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα περνάμε στους ομιλητές από τις πολιτικές ομάδες για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για πέντε λεπτά το λόγο έχει ο Γιώζεφ Σάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο λέμε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη περίοδο της ιστορίας της και την τρέχουσα εβδομάδα νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι αυτό ισχύει. Αλλά αυτό υπογραμμίζει όλα όσα είπαμε για την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της Ένωσης. Η άσκηση συζήτηση του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι παρόμοιο. Ας δούμε τι έχει γίνει πριν από κάποιο καιρό και χαίρομαι που ο Αντιπρόεδρος ξεκίνησε με μια απαρίθμηση των όσων έχουν ήδη γίνει, γιατί είδαμε κι εμείς και παρατηρήσαμε και παρακολουθήσαμε τα όσα συμβαίνουν. Θα έλεγα από πλευρά του ΕΛΚ ότι μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια γρήγορη και καλή αρχή το επενδυτικό πακέτο, πολλέ άλλε πρωτοβουλίε πολύ ισχυρέ. Και εμεί από πλευρά του Κοινοβουλίου θα θέλαμε να βοηθήσουμε στην διαδικασία αυτή για να προχωρήσουμε στους τομείς αυτούς. Και θα πρέπει λοιπόν αυτή η δυναμική αρχή να συνεχιστεί. Θα θέλαμε επίση να σχολιάσουμε το εξή. Ένα πράγμα που πολλοί έχουν παραμεινεύσει, την απόφαση του Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου σε ό,τι αφορά για την έλλειψη υποστήριξη σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της ε, εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Κανονικά σε χρόνια, σε έτη ε, εκλογών δεν σε κάτι τέτοιο γιατί χρειάζεται πολύ πιο πολύ χρόνο. Δεν ε, μπορούμε να τα προετοιμάσουμε όλα αυτά. Φέτος όμως μπορούμε να τα προετοιμάσουμε αυτά. Προφανώς δεν ε, αν λέω ότι είναι τέλεια η διαδικασία προπαρασκευής. Στις διαπραγματεύσεις που γίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο συζητήσαμε όλα όσα έγιναν το τελευταίο μισό έτος, όλους τους συμβιβασμού που προβλέπουμε για το επόμενο έτος, για το δεύτερο ημίση του τρέχοντος έτους, αυτό είναι πολύ βαρύ και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τους ίδιους διαπραγματεύσεις, τις ίδιες συμβιβασμούς. Ωστόσο, ασκώντας μια πολύ σημαντική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, η πρωτοβουλία της ανάληψης πρωτοβουλίας, έχουμε δύο εργαλεία, δύο μέσα για να πετύχουμε κάποιες ιδέες ε, και να τις προβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναμένουμε δε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις αυτές. Χαίρομαι που ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι θέλουμε αποτελεσματική νομοθεσία να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία, σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού άχθους λοιπόν, μεταφορά, εφαρμογή τη ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ε, πολύ συχνά δεν χρειάζεται κανένα ε, νομοθεσία, πολύ απλά χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά η ήδη υφιστάμενη νομοθεσία. προφανω δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα ματαιοδοξία για το ποιο θα πάρει την έκθεση ή την νομοθετική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο εντελεχείς εδώ στο Κοινοβούλιο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε θέματα εφαρμογής. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό λοιπόν πλήρω υποστηρίζουμε την καλύτερη διαδικασία κατάρτισης νομοθεσίας. Επίσης, η εναρμόνιση της νομοθεσίας ε, στην συνθήκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις. Μεγάλη καθυστέρηση και μεγάλη αντίρρηση και μεγάλη... Μεγάλος δισταγμός από πλευράς ε, του Συμβουλίου. Θα πρέπει να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πλήρη δικαιώματα για να μην έχουμε διαρκώς διαθεσμικές διαφωνίες, να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Είναι πραγματικά αδύνατο το γεγονός ότι δεν το έχουμε ήδη πράξει. Και δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποσύρει την νομοθεσία αυτή. Ελπίζουμε ότι η καλύτερη νομοθεσία και στο πακέτο αυτό θα συμπεριληφθούν ε, και άλλε προσπάθειε προ την κατεύθυνση αυτή. Ε, θεωρούμε ότι οι θέσει απασχόληση παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα. Η ευελιξία, η κινητικότητα, η απασχόληση των νέων, η ψηφιακή ατζέντα παίζει σημαντικό και θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μα. ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αναζήτηση θέσεων εργασία, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση τη νέα γενιά, την καλύτερη πρόσβαση στι ψηφιακέ υπηρεσίε στην επόμενη εξέλιξη της Νομισματικής Ένωσης θα πρέπει να βασιστεί στην νομοθεσία 2-pack και 6-pack, δέσμης 2 και 6 οδηγιών. Θέλουμε αυτά τα δύο εργαλεία να εφαρμοστούν πλήρως για την πολιτική φορολόγηση που αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της μεταρρύθμισης των κρατών μελών. Θα θέλαμε να δούμε εξελίξεις, να μεταφερθεί η φορολογία από τη φορολογία εργασία σε άλλου είδους φορολογία σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, η καταπολέμηση τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, η υποστήριξη καλύτερη απόδοση του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού αποτελούν σημαντικά ζητήματα. Σε γενικέ γραμμέ, για να συνοψίσω, θα θέλαμε τώρα το Κοινοβούλιο να βγει και να πει ότι θέλουμε κι εμεί να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή. Και αυτό ελπίζουμε ότι θα πετύχει το ψήφισμά μας. Ελπίζω ότι οι πολλοί συνάδελφοι εδώ στο Κοινοβούλιο θα υποστηρίξουν τα κοινά ψηφίσματα τα οποία και προετοιμάσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Για τους Σοσιαλιστέ και δημοκράτες, το λόγο έχει ο Ρίκε Γκρέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για μία διπλή άσκηση. Αφενός έχουμε και πρέπει να καταγράψουμε το τι έχει συμβεί από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από, από το πρόγραμμα το οποίο μα παρουσίασαν στην αρχή. Και επίση θα πρέπει να δοθεί μια δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεισφέρει στην ε, κατεύθυνση που θέλει να δρομολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι τμήμα τη διαθεσμική συμφωνία. Αλλά νομίζω ότι ξεπερνάει και τα όρια μια συμφωνία, λόγω του ότι έχει υψηλότατη πολιτική σημασία. Γι' αυτό ακριβώ το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι τμήμα αυτή τη πολιτική κατεύθυνση που παίρνει η Ένωση. Όταν προσπαθούμε να δούμε τι συνέβη σε αυτό το πρώτο τμήμα τη ε, δράση τη Κομισιόν, η αξιολόγηση που κάνω είναι πραγματικά θετική. Το μείγμα του προγράμματος επενδύσεων Η ευελιξία του προγράμματος ανάπτυξης επέτρεψε να δοθεί μια νέα τροπή στην οικονομική πολιτική της Ένωσης και να, και να κατευθυνθεί προς τα ε, στοιχεία που χρειάζονται να λάβουμε υπόψη μας. Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτά είναι που πρέπει να δούμε τώρα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Η Κομισιόν μας κάνει μια ουσιαστική ε, πρόταση για τα φορολογικά θέματα και επίσης κάνει και μια σημαντικότατη και αξίαπαινη πρόταση για την ε, μετανάστευση. Και οι θέσεις της είναι φιλόδοξες για την ενεργειακή πολιτική, καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν την οικονομική πολιτική. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η διαφάνεια υπάρχει στη συμπεριφορά της Κομισιόν, το βλέπουμε και αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο. Αντιμετωπίζουμε τώρα τι προκλήσει του 2016. Εμεί έχουμε συγκεκριμένε προτεραιότητε, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό πεδίο, σε ό,τι αφορά το θέμα τη μετανάστευση και σε ό,τι αφορά τη φορολογική πολιτική και στο, σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα θα θέλαμε όλε οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι οριζόντιε και να οι πολιτικέ να διέπονται από μια κοινωνική διάσταση. Αυτά θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα θέματα. Δεν αρκεί να πούμε ότι είμαστε υπέρ μια κοινωνική πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχει και κάτι το απτό. Μπορούμε να συνεργαστούμε ούτω ώστε να δώσουμε σάρκα και οστά στα στοιχεία που αφορούν την ε, καταπολέμηση της στόχια, του, της στόχιας, του αποκλεισμού, ε, το σεβασμό των συλλογικών ε, συμβάσεων. Όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος μόλις τώρα, μόλις τελειώσαμε την νομοθεσία για την κινητικότητα των εργαζομένων και τα δικαιώματά τους στα πλαίσια αυτής της κινητικότητας. Είπατε ότι θα παρουσιάσετε ένα πακέτο για την ΟΝΕ επίσης. Και στα πλαίσια της ΟΝΕ θα θέλαμε το κοινωνικό στοιχείο, την κοινωνική διάσταση να την καταστήσουμε βασικό στοιχείο της ΟΝΕ. της ενισχυμένης αυτής και αναθεωρημένης ΟΝΕ. Όχι μόνο στο κείμενο των Προέδρων, αλλά σε όλε τι δράσεις που προωθεί η Κομισιόν. Φορολογική πολιτική. την πρόταση μπορούμε να την και να πούμε ότι έχει δύο πτυχές. Θα θέλαμε να αφορά να εστιάσουμε στις χώρες όπου δημιουργούνται τα κέρδη. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή φορολογική εταιρική βάση. Στο θέμα της μετανάστευσης, αυτό που επιθυμώ είναι η Κομισιόν να διατηρήσει την ορμή που παρατηρήσαμε μέχρι τώρα και να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να αναλάβουν αλληλέγγυα τα βάρη τους. Ε, βάρη που δημιουργούνται λόγω της ανθρωπιστικής ε, κρίσης. Και πιο μακροπρόθεσμα να μας κάνει προτάσεις για να οργανώσουμε σοβαρά την ε, νόμιμη μετανάστευση και να την πλαισιώσουμε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιμετωπίσουμε με αλληλεγγύη το θέμα του ασύλου. Και κλείνοντας θα μιλήσω για τη δημοκρατία. Θα ήθελα, η ομάδα μου θα ήθελε, να παρουσιαστεί μια πρόταση με δείκτες αντικειμενικούς και με ένα υποχρεωτικό μηχανισμό για να απαντήσουμε στις ρογμές και στις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης. Και αυτά θα πρέπει να υπάρχουν στις συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Next speaker, on behalf of the European... Από πλευρά των συντριστών και μεταρρυθμιστών, ήδη ε, για δύο λεπτά η κυρία Βίκη Φόρντ. Ευχαριστώ. Πέρσι, εδώ ακριβώς, ε, μιλούσαμε για ε, προκλήσεις ανεφροηγουμένου για την οικονομία, για τους πόρους και για την ασφάλεια μας. Και σήμερα στην Ευρώπη δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση και το αντίθετο έχει επιδεινωθεί σε πολλέ χώρε. Χρειάζεται αλλαγή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, αυτή η μόνιμη πορεία προς την ε, ε, ε, ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι λύση και δεν το υποστηρίζουμε. Όσα χρόνια είμαι εγώ εδώ ζούμε μια ε, σοβαρή οικονομική κρίση και βλέπουμε όμως ότι η δική μας οικονομία στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει τις περισσότερες θέσεις εργασίας χάρη στο μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό και έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη περισσότερες θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να νομοθετεί διαρκώ χωρί να εξετάζει τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα νέα νομοθετήματα θα πρέπει ταυτόχρονα να ε, μεριμνά ούτω ώστε να μην συνιστά με μεγάλο άχθο και απαράδεκτη γραφειοκρατία για τι επιχειρήσει, ήδη υφιστάμενη νομοθεσία. Οπότε θα πρέπει αυτό το απλό καθήκον να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όταν είναι να νομοθετήσει, να εξετάζει αν θα είναι ευκολότερη ή δυσκολότερη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, ε, η ενιαία αγορά τι νόημα έχει να είναι ευχερέστερες οι εμπορικές συναλλαγές. Ε, το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με την ψηφιακή οικονομία. Δηλαδή να υποστηρίξουμε την ψηφιακή επανάσταση, όχι να την υπονομεύσουμε. Και σε αυτή την έκθεση το βλέπουμε ξεκάθαρο αυτό. Επίσης πρέπει να υποστηρίξουμε τις εμπορικές συναλλαγές. Ε, ναι, ας εφαρμόσουμε τη συμφωνία με τον Καναδά και ας συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε με τις ΥΠΑ. Χρειαζόμαστε επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα διότι είναι οξύτερη η κρίση του δημοσίου χρέους σε σχέση με το παρελθόν. Χρειαζόμαστε αυτέ τι επενδύσει και πρέπει να σταματήσουμε να ισχυριζόμαστε ότι είναι ίδια όλα τα δημόσια χρέη και ε, έχουν κέριο ρόλο οι διαρθωτικέ αλλαγέ. Δεν έχουμε περιθώριο ελίγμων, ε, διότι ε, χρειαζόμαστε λίγο μικρότερη, πιο περιορισμένη νομοθεσία, πολύ εστιασμένη νομοθεσία, ούτω ώστε να υπάρξει διακομματική υποστήριξη. Θα μπορούσαμε να σε υποστηρίξουμε αν αναδείξετε σε προτεραιότητα την ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεργαστούμε με όσου μοιράζονται αυτό το όραμα. Σα ευχαριστούμε κυρία Φόρδα από πλευρά των φιλελευθέρων. Τρία λεπτά η Σοφή Ιντβέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε χαμογελάσετε ίσως για το ότι το ψήφισμα του Κοινοβουλίου ξεκινάει λέγοντας ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε στα μεγάλα και μετά μα χρειάζονται 29 σελίδε για άλλα πράγματα, τα σημαντικά, τα ουσιώδη. Καλωσορίζω ιδιαίτερο τον στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που υποστηρίζεται από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Πάντα είναι σωστό και καλή ιδέα αυτό παντού. Αλλά δεν θα πρέπει να καταστεί αυτό, αυτό, σκοπό και να σα πω με πάσα ειλικρίνεια, η μείωση τη γραφειοκρατία δεν αποτελεί την απάντηση στι μεγάλε προκλήσει τη σημερινή, δεν αποτελεί την απάντηση στο θέμα των προσφύγων, τη κρίση τη Ευρωζώνη, δεν είναι η απάντηση για την ε, κατάρρευση τη ε, ε, ζώνη Σέγγεν, τη κρίση με τον Πούτιν. Χρειαζόμαστε λοιπόν και πιο πολλά πέρα από τη μείωση τη γραφειοκρατία και να θυμόμαστε ότι αυτά που κάνουμε εδώ σήμερα είναι πράξεις για την ίδρυση και την εγκαθίδρυση, την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία θα ζήσουν οι μελλοντικές γενιές. Για αυτές δουλεύουμε, για τις μελλοντικές γενιές. Μία πρώτη παρατήρηση για την καλύτερη νομοθεσία. Για μένα πρόκειται πιο πολύ για μια διαδικασία, όχι τόσο για ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι θέμα πολιτικής απόφασης και στη διαδικασία αυτή πολλά πρέπει και μπορούν να βελτιωθούν. Και εδώ μπορεί να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή μιας πραγματικής κουλτούρας διαφάνειας και πρόσβαση στα έγγραφα, γιατί παρά όλες τις όμορφες κουβέντες, θεωρώ ότι οι τρεις θεσμοί, και αυτό περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξακολουθούν να έχουν πολύ συντηρητικέ ε, αντιδράσεις σε ό,τι αφορά την διαφάνεια. Δεύτερο και ίσονο σημασία, δεν περιλαμβάνεται στο ψήφισμα, αλλά νομίζω ότι εκπροσωπεί τους πιο πολλούς, όλους δηλαδή, είναι να έχουμε σαφείς, πραγματικές και σοβαρές απαντήσεις Στι κοινοβουλευτικές μας ερωτήσεις και όχι αυτές τις ε, εικονικές απαντήσεις που λαμβάνουμε. Επίσης, να αντιδρούμε στις νομοθετικές προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εσείς, κύριε Επίτροπε, δηλώσατε ότι πρόκειται να το κάνετε αυτό, γιατί είναι πραγματικά περίεργο. Μια πρωτοβουλία πολιτών που περιλαμβάνει και προϋποθέτει ένα εκατομμύριο υπογραφές να υποχρεώνει την Επιτροπή να απαντήσει αλλά αυτό το κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τόσα εκατομμύρια εκλογής ε, που ψήφισαν πέρσι να αγνοείται. Μπορεί λοιπόν να τα πάει πολύ καλύτερα σε θέματα ε, και αναθεώρησης και αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλο για αυτά τα μεγάλα πράγματα τα οποία συζητάμε συγκαταλέγεται και η βελτίωση των, της Ευρωζώνης και αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο την Ελλάδα αλλά θα πρέπει να πάμε πιο πέρα από την πρόταση των πέντε προέδρων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να συνταχθούν για την κατάρρευση της ζώνης Σέγγεν. Και τέλος, αν μου επιτρέπετε πρόεδρε να κλείσω το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει ένα μηχανισμό για την εφαρμογή του άρθρου 2 για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτο δικαίου. Αυτό πιστεύω ότι και ελπίζω να, του δώσω σημασία, να δώσω σημασία η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια για την Ηνωμένη Αριστερά, δύο λεπτά η Κριστίνα Ζούμπερ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όπου διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι λαοί του βιώνουν ε, δραματικές στιγμές που θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο την καθημερινή του ζωή των πολιτών, των ε, εργαζομένων αλλά και το μέλλον ε, των χωρών πρέπει να γίνει η ρήξη με τις παρελθούσες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι θεωρούμε ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου των χρηματοπιστωτικών αγορών. Θα καταθέσουμε λοιπόν πρόταση και τροπολογίες σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ε, χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα η σημερινή πολιτική για να συνεχιστούν οι τωρινές πολιτικές. Ε, ε, πρέπει να αλλάξει η σημερινή πολιτική ούτως ώστε η ανάπτυξη να φτάσει σε βιώσιμο επίπεδο και να ε, υπάρχουν χρέη που μπορούν να αποπληρωθούν. Για το Σύμφωνο Σταθερότητας και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο θα προτείνουμε τροπολογίες ε, εν ώψη και της αναθεώρησης ε, της πολιτικής για την ΟΝΕ και θα προτείνουμε και ειδικέ ρυθμίσεις που θα προσαρμόζονται στις ειδικέ ανάγκες σε κάθε χώρα. Πρέπει να αντικατασταθεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο με ένα σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση υπέρ όλων των χωρών. Θα προτείνουμε μια διακυβερνητική διάσκεψη με στόχο να τροποποιηθεί και να αντικατασταθεί το Δημοσιονομικό Σύμφωνο. Χρειάζεται επίσης ε, με τροποποίηση της εντολής ε, και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να αυξήσουμε τον πολιτικό έλεγχο ε, της δραστηριότητάς του και να μειώσουμε την επιρροή από τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για θεμελιώδη ζητήματα για τα οποία παίρνει αποφάση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που σχετίζονται με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και γι' αυτό χρειάζεται η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας νομοθεσία. Επίση, χρειάζεται τροποποίηση νομοθεσία για την Τραπεζική Ένωση. Δεν είναι βιώσιμο πλέον το τραπεζικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε επιτέλου τα συμφέροντα των πολιτών και των εργαζομένων. Η πολιτική δεν θα πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, τα συμφέροντα των πολιτών. Με τι ε, τροπολογίε μα θα ξεκαθαρίσουμε τι θέσει πολιτικέ μα ομάδα σε αυτά τα κεντρικά ζητήματα. Για δυόμιση λεπτά από τους πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την εισαγωγή της. Καταρχά όλοι μα μπορούμε να συμφωνήσουμε επί ενό πράγματος, ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι φιλόδοξη για τα μεγάλα πράγματα και ταπεινή για τα μικρά. Το θέμα είναι ποια είναι τα σημαντικά και φιλόδοξα και ποια είναι τα πιο ασήμαντα. Και αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση και πολιτική απόφαση. Και α μην κρυβόμαστε πίσω από μελέτε αντικτύπου ή πίνακε ελεγκτικούς. Πρέπει να γίνει μια πολιτική συζήτηση για το τι είναι μεγάλο και τι είναι μικρό και όπου θέλουμε, πού θέλουμε να βάλουμε την Ευρώπη μπροστά, να την προτάξουμε. Υπάρχουν πολλές επικρίξεις ε, για το πώς δουλεύει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν πολλοί κανόνες ε, που θεσπίζουν οι Βρυξέλλες ή γιατί λόγω της κατάστασης στην Ελλάδα. Λόγω της αυξανόμενης ανεργίας στην Ευρώπη ή λόγω της ε, αυξανόμενης ανισότητας. Το δεύτερο νομίζω η Ευρώπη θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει τις ανισότητες και που γίνεται πιο κοινωνική, πιο βιώσιμη. Και αυτά είναι τα σημαντικά πράγματα, αυτά είναι τα μεγάλα πράγματα, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση της Ευρώπης. Και εκεί θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κύριε Τίμερμανς, είπε, είπατε, ας ξεφορτωθούμε το μύθο ότι αυτή η Κομισιόν δεν είναι προοδευτική, ότι δεν είναι φιλόδοξη και δεν νομοθετεί αρκετά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι πρέπει να μας δώσετε κάποιες αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Ε, και αυτό θα αποδειχθεί όταν μας προτείνετε τις πιο φιλόδοξες προτάσεις, όπως λέτε, για την κυκλική οικονομία. Θέλουμε να δούμε ποιε είναι αυτές οι πιο φιλόδοξες. Είπατε στην ομάδα μου ότι θα μας διαψεύσετε, επειδή ήμασταν ε, λίγο σκεπτικιστέ. Αλλά πρέπει να μου το αποδείξετε. Το ίδιο και για τη μετανάστευση και για το πρώτο ε, σχέδιο με την της Κομισιόν, που ήταν καλό, το υποστηρίξαμε. Αλλά ξέρετε ότι αυτό είναι μόνο η απαρχή μια μεγάλη συζήτηση. Και εδώ η Κομισιόν θα πρέπει να πει τι πιστεύει. Ε, Πώ θα μπορούμε, α πούμε, για την νόμιμη μετανάστευση να δημιουργήσουμε νόμιμε οδού πρόσβαση. Το ίδιο για τη φορολογία. Η φορολογία, το πακέτο φορολογία μέχρι στιγμή δεν είναι πολύ φιλόδοξο. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και αναχώρα ε, υποβολή εκθέσεων. Επίσης, για την ονέα λέτε ότι πρέπει να είναι πιο ε, δημοκρατική και πιο κοινωνική. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα συζητήσουμε και τελικά όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε μαζί. Περιμένουμε να συνεργαστούμε λοιπόν ε, με βάση την διαθεσμική συμφωνία. Αλλά επίσης όρις και ας μην κρυβόμαστε πίσω από ευρωκρατικές μελέτες αντικτύπου. Ας κάνουμε πραγματική πολιτική συζήτηση και όλα τα, τρι... τα θεσμικά όργανα, τα τρία βασικά θεσμικά όργανα, να είναι στο ίδιο επίπεδο. Ο επόμενο ομιλητή. Από το EFTD, ε, ο κύριος Μπορέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από όλα όσα συνέβησαν αυτή τη βδομάδα, την περασμένη, την Κυρία που μας πέρασε στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως πριν. Συνέβη κάτι τρομερό κάτι που πρέπει να μας κάνει όλοι να αναλάβουμε τις ε, θεσμικές μας ευθύνες και πρέπει να μάθουμε. Το μήνυμα που μας έστειλε η Αθήνα δεν ήταν τεχνικής φύσεως που αφορά μόνο το θέμα της ε, ερώτησης, αλλά είναι και πολιτικό το μήνυμα. Ε, όλα τα πολιτικά θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο που είναι η άμεση έκφραση της ε, βούλησης των πολιτών πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το πολιτικό νόημα που είχε αυτό το μήνυμα. Θα πρέπει η Κομισιόν Γιούνκερ να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη τα σημαντικά δρόμενα της περασμένης εβδομάδα. Θα πρέπει η Κομισιόν πραγματικά να δείξει αυτή την πολιτική πρωτοβουλία με χρήσιμες προτάσεις για όλους τους λαούς της Ένωσης και κυρίως απέναντι στους πιο ευπαθείς. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε το σχέδιο Juncker με βάση κριτήρια που θα λαμβάνουν υπόψη γεωγραφικές περιοχές που έχουν περισσότερες δυσκολίες. Πέρα από την αξία ή τις ε, ευθύνε που έχουν οι κυβερνήσεις, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει στο κέντρο των σκέψεών μας να έχουμε τους λαούς. Η Κομισιόν έχει ε, τον έλεγχο της ε, πολιτικής πρωτοβουλίας. Το χρησιμοποιεί με προσοχή και σύνεση και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αλλά και με αλληλεγγύη. Τα επιμέρους μέτρα θα πρέπει, κατά την άποψή μας, να επικεντρωθούν κυρίως στην ε, υψηλή ανεργία, ε, σε μία αύξηση που δεν την βλέπουμε, σε υψηλά ε, επίπεδα χρέους, σε ένα σύστημα πιστοτικό το οποίο δεν λαμβάνει την κατάσταση υπόψη την κατάσταση των οικογενειών και των επιχειρήσεων και μια πολιτική μετανάστευση και καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν κάποια εγκάρσια δεινά. Διαφθορά, φοροδιαφυγή, ε, διήθηση του, στο, του οργανωμένου εγκλήματος στην πραγματική ζωή που απαιτούν σε κοινωνικό επίπεδο μια πιο συγκεκριμένη και στοχοθετημένη δράση. Δεν μπορούμε εμείς να επιτρέψουμε να ε, αφήσουμε τους πολίτες να χάσουν την εμπιστοσύνη τους σε εμάς. Η Κομισιόν με το πρόγραμμα εργασίας της μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Μπορούμε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας από τους ε, εκλογείς μας. Ελπίζουμε και θέλουμε να κάνει καλά τη δουλειά της η Κομισιόν και να την κάνει κυρίως με ευσυνειδησία. Σας ευχαριστώ και κυρίως που τηρήσατε και το χρονικό όριο. δύο λεπτά από την Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας, ε, ο κύριος Φοντάνα. Πάρα πολλά πράγματα έχω να πω σε αυτή τη συζήτηση, Επίτροπε. Η εντύπωση που έχω σήμερα είναι ότι σε κάνα χρόνο θα ξαναβρεθούμε εδώ και θα λέμε τα ίδια και η κατάσταση θα είναι και χειρότερη μάλιστα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι θέλει να κάνει η Κομισιόν. Όχι μόνο για το μέλλον τη, αλλά για το μέλλον τη Ευρώπη. Τουλάχιστον για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πραγματικά δεν καταλαβαίνω εάν η Κομισιόν συνειδητοποιεί ότι παίρνει όλο και μεγαλύτερους, λαμβάνει όλο και μεγαλύτερους κολάφους. Πρέπει να κάνουμε, για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, ε, πρέπει να κάνουμε δράσεις, να προωθήσουμε δράσεις πολύ στοχοθετημένες και αποφασιστικές για να ξαναβρούμε την ε, ευημερία. Γιατί αντί για την ευημερία βλέπουμε ε, την καταστροφή κάποιων λαών. Το μήνυμα που έστειλε η Ελλάδα τη περασμένη εβδομάδα είναι πολιτικό μήνυμα και σα παρακαλώ, σα κάνω έκκληση, σα εκλυπαρώ να αλλάξετε την πολιτική, ε, την πολιτική σας. Γιατί το σχέδιο Juncker που προβλέφθηκε πέρυσι δεν αρκεί. Πάνω απ' όλα όμως θα πρέπει να μας εξηγήσετε ποιες είναι οι πραγματικές σας προτεραιότητες. Ίσως δεν λέγονται αυτές οι πραγματικές προτεραιότητες. Εμεί έχουμε στο μυαλό μα τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, τι παραδόσεις μα, την ταυτότητά μα. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη είναι δυνατή γιατί είναι διαφορετική. Αντίθετα, εσεί προωθείτε πολιτικέ δράσει που έχουν σαν στόχο τι πολυεθνικέ και τι μεγάλε τράπεζε. και όλου αντιμετωπίζετε σαν νούμερα. Αυτό δεν το δεχόμαστε. Και βλέπετε ότι οι λαοί εξεγείρονται. Σκεφτείτε ότι το made in, η οδηγία για το made in είναι μπλοκαρισμένη. Και ενώ προχωράτε ας πούμε για το TTIP που όλοι πολύ καλά ξέρουμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποιε μεγάλε πολυεθνικέ, αλλά δεν θα είναι χρήσιμο για τι ε, μικρέ εταιρείε μα, τουλάχιστον έτσι φαίνεται, εσεί δεν κάνετε τίποτα πέραν του TTIP. Επίση, ποια είναι η ματιά μας για τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα για τους ε, χριστιανούς αδερφούς μας που διώκονται. Εδώ μιλάμε για φοβίες, ισλαμοφοβίες κτλ. Αλλά δεν μιλάμε καθόλου για την χριστιανοφοβία. Και για το Ισλαμικό κράτος τι λέμε. Μία δράση στοχευμένη της Ευρώπης για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας απέναντι στο μεγαλύτερο κίνδυνο που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Τι κάνουμε γι' αυτό. Η κυρία Κριστίνα Μόρβα έχει το λόγο ως ε, Το νέο πρόγραμμα εργασία ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δηλώνει με πάσα σαφήνεια ότι υποστηρίζει όλε τι νόμιμε μορφέ μετανάστευση και θα χρησιμοποιήσει μάλιστα σκληρά μέτρα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό λοιπόν το παρέθεσα. Ρωτώ λοιπόν αγαπητέ Επίτροπε, θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε Ποια είναι η διαφορά, τι είναι η νόμιμη και παράνομη μετανάστευση. Ξέρουμε ότι η νόμιμη μετανάστευση είναι κάποιος που ζητά το καθεστώς πρόσφυγα γιατί θέλει να διαφύγει από τον πόλεμο στην πατρίδα του. Γιατί όμως ένα τέτοιο άτομο θα πέταγε τα διαβατήριά του στα σερβικά ουγγρικά σύνορα. Γιατί δεν δηλώνει ότι είμαι από τη Συρία όπου επικρατεί πόλεμο. Σας παρακαλώ να γνωρίσετε το καθεστώς του πρόσφυγα που κατέχω και ειδού και τα έγγραφά μου. Αν ναι, φεύγουν και διαφεύγουν από τον πόλεμο, πώς είναι δυνατόν να αφήνουν τα γυναικόπαιδα πίσω τους. Ε, μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτά. Και έτσι λοιπόν ε, ολοκληρώθηκε ο κύριος ε, των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων και των μεν εγγεγραμμένων. Και το λόγο έχει τώρα ο κύριο Τίμερμαν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε μια σειρά σχολείων που έγιναν. Καταρχά, να πω ότι υπάρχει ευρεία υποστηρίξη για την πιο στενή συνεργασία και το πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι στοχευμένο. Και ασφαλώς θα πρέπει να τεθούν πολιτικές προτεραιότητες και θα πρέπει να συζητηθούν αυτές οι πολιτικές προτεραιότητες για να υποστηριχθούν από την πλειοψηφία. Εκ παραλίλου βλέπω προθυμία από το Κοινοβούλιο, όπως ξέρω ότι πίσταται προθυμία και στο Συμβούλιο και ε, στην Επιτροπή για να Υπάρχει διαθεσμική συμφωνία μέχρι τα τέλη του έτους, ελπίζουμε, για την καλύτερη νομοθεσία. Και φυσικά η καλύτερη νομοθεσία δεν απαντά την απάντηση σε όλα τα προβλήματά μας. Δεν πρόκειται να επιλύσει την κρίση στην Ελλάδα. Η καλύτερη νομοθεσία ούτε αποτελεί την απάντηση στα προβλήματα του Πούτιν. Τα αποδέχομαι αυτά. Όχι όμως, αποτελεί ένα καλό τρόπο να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στην έκκληση ε, ατελείωτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη όποτε επισκέπτομαι κάποιο κρατός που μας λένε σας παρακαλώ λίγη σαφήνεια, λίγο λιγότερη γραφειοκρατία, σας παρακαλούμε βοηθέστε μας να κατανοούμε την νομοθεσία, να μην υπάρχει νομοθεσία που να είναι ανοιχτή σε ατελείωτες ε, ερμηνείες από τα κρατημέλη. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι σημαντικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικές και για την απασχόληση και για την ανάπτυξη με τη σειρά της. Και ασφαλώς αυτό δεν αποτελεί κάτι το οποίο θα αλλάξει την φύση της Ευρώπης. Θα κάνει όμως μια διαφορά για εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που καθημερινά, κάθε μέρα εργάζονται σκληρά για να βγάλουν το ψωμί της οικογένειάς τους και για να συντηρήσουν τους εργαζόμενους τους. Γι' αυτό λοιπόν αυτό μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο. Ο τρόπος που τον οποίο καταρτίζουμε νομοθεσία είναι σημαντικός για εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια μάλιστα Ευρωπαίους, ακόμα και αν δεν το ξέρουν. Εξακολουθεί να είναι βασικό, γιατί το αποτέλεσμα είναι κάτι με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι. Και να είμαι και λίγο ξεκάθαρο τα θέματα μελετή αντικτύπου. Και για την αύξηση του ελέγχου. Αυτό δεν σημαίνει ότι παίρνουμε την εξουσία από τα χέρια των πολιτικών. Όχι. Θα μας οδηγήσει σε πιο καλά ενημερωμένους πολιτικούς. Και εδώ δεν βλέπω ποιο είναι το πρόβλημα. Καλύτερος έλεγχος, καλύτερες μελέτες αντικτύπου. Αυτό τι σημαίνει, ότι όταν θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις οι πολιτικοί θα είναι πιο καλά ενήμεροι γι' αυτό στο οποίο θα πρέπει να αποφασίσουν. Και θα ήθελα να σας πω να μην αντιστρέφουμε τα επιχειρήματα ότι η πολιτική θα πρέπει να είναι ε, αυτοί που κινούν τα νήματα και γι' αυτό λοιπόν απορρίπτουμε την ε, παρακολούθηση, απορρίπτουμε όλη αυτή την ενημέρωση και τις μέρες του αντικτύπου. Όχι, δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά για να σας πάρουμε τη δύναμη. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους πολιτικούς να είναι πιο καλά ενημερωμένοι και το βλέπουμε σε όλα τα κρατημέρια ότι κάποιες φορές ο, ο έλεγχος, η ανάλυση, η παρακολούθηση οδηγούν σε κάποια απορίσματα για το κόστος, για παράδειγμα, των μέτρων και μετά παρόλα αυτά τα κοινοβούλια αποφασίσουν ότι πιστεύουμε ότι δικαιολογείται αυτό το μεγαλύτερο κόστος αλλά τουλάχιστον ξέρουμε τι αποφασίζουμε. Και αυτό νομίζω ότι είναι προφανές και απαραίτητο για την πιο πολύ διαφάνεια τώρα. Είμαι υπέρ. Και ένας από τους λόγους για τον οποίο χρειαζόμαστε εμείς τα διαθεσμικά όργανα πιο πολύ διαφάνεια είναι για να δείξουμε μεταξύ άλλων στους πελάτες μας, στους αποδέκτες της νομοθεσίας μας, που είμαστε εμείς υπεύθυνοι, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και που είναι αρμόδιοι, οι εθνικές κυβερνήσεις και γιατί εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη παρανόηση. Και πάλι τα κράτη-μέλη έχουν την ε, αρμοδιότητα να το πράξουν. Αν θέλουν να είναι πιο αυστηροί σε κάποιου τομεί, έχουν απόλυτο δικαίωμα να το πράξουν. Αλλά να είναι τουλάχιστον ειλικρινεί, να μην τα ρίχνουν όλα στις, ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και έτσι απαντάω και στον κύριο Ζάιρ και για τι πράξει κατά εξουσιοδότηση και τι εκτελεστικέ πράξει. Ε, ελπίζω να πετύχουμε μια συμφωνία για πιο πολλή διαφάνεια από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα σχέδια πράξεων κατά θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για περίοδο 4 εβδομάδων για να, να βλέπουν όλοι τι προτείνεται. Οι εκτελεστικέ πράξει είναι λίγο πιο δύσκολε. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για την αλλαγή μια τιμή, δεν μπορούμε να το δώσουμε αυτό στη δημοσιότητα. Αυτό το καταλαβαίνουν όλοι, νομίζω. Αλλά η πρωτογενή και η νομοθεσία θα δημοσιεύονται και ελπίζουμε έτσι να καταφέρουμε να πετύχουμε την ε, επόμενη πιθανή καταστροφή. Και φυσικά θα πρέπει να δράσουμε για μια σειρά ε, ζητημάτων. Η μετανάστευση είναι ένα θέμα εξ αυτών. Είμαι σίγουρος ότι αύριο όταν θα γίνουν ε, συζητήσεις για τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Γιούγκροφ θα συζητήσει αυτό και πιστεύουμε ότι είμαστε στη σωστό δρόμο στο διαφορά τις προτάσεις αυτές και να σας πω ότι αν μας ρωτάτε τι είναι η διαφορά μεταξύ της νόμιμης και της παράνομης μετανάστευσης, κάποιος που συστήμα του συστήματο ασύλου γιατί θέλει μια πιο καλή ζωή στην Ευρώπη, αυτό αποτελεί παράνομη μετανάστευση. Και οι τον άσυλο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ε, φύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους. Πολλοί από τους πολίτες μας γνωρίζουν ότι το σύστημα είναι ανοιχτό σε καταχρήσεις και δεν ε, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να επιστραφούν όλοι ότι επιστρέφονται τα άτομα που πρέπει να επιστρέφουν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι εφαρμόζονται οι κανόνες προκειμένου όσοι αξίζουν το άσυλο το λαμβάνουν και δυστυχώς το σύστημα συχνά αποτυγχάνει ενώ όσοι δεν ε, ε, δικαιούνται άσυλο θα επιστρέφονται και υπάρχουν συμφωνίε με τρίτε χώρε για να συμβαίνει αυτό αλλά αυτό που χρειαζόμαστε και αυτό αποτελεί απλά δημογραφική πραγματικότητα θα πρέπει να υπάρχουν ε, δυνατότητε παραδοσιακή, νόμιμη μορφή μετανάστευση στην Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να ζητά κανεί μια θεώρηση στην πρεσβεία του και να έρθει να δουλέψει και να ζήσει στην Ευρώπη. Όχι να είναι στο έλεο των διακινητών και να Ρίσκαρ τη ζωή του στη Μεσόγειο. Η Ευρώπη λοιπόν χρειάζεται τέτοια άτομα που ενδεχομένω θα κάνουν έτσι να έρθουν στην ε, Ευρώπη. Άρα και θεωρώ ότι η νόμιμη μετανάστευση αποτελεί μέρο τη λύση. Και θα ήθελα να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, διευκρινίζοντα το εξή, ότι για μένα το σημαντικό είναι ότι τα διατασμικά όργανα, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, θα συνεργαστούν στενά. Γιατί νομίζω κανεί δεν ε, αμφισβητεί τον στόχο ότι θα πρέπει να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα για του πολίτε μα. Κάποιες ε, φορές τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, αλλά σε διάφορες περιστάσεις ε, είναι μικρά και ανεπαίσθητα τα αποτελέσματα, τα οποία όμως δημιουργούν καλύτερη ανάπτυξη, καλύτερες θέσεις εργασίας, καλύτερη επιχειρηματικότητα, καλύτερη... καλύτερες θέσεις εργασίας για τους ε, εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους σήμερα στην Ευρώπη. Αυτός πιστεύω είναι ένας στόχος που αξίζει τον κόπο να τον επιδιώξουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιπρόεδρο Τίμερμαντς. Επτά ψηφίσματα έχουν καταδεθεί. Κλείνει η συζήτηση.